Καλημέρα σε όλους. Παρακαλώ, πάτε τις θέσεις σας. Κάντε και λίγο ησυχία, αν γίνεται. Καλή σας μέρα. Υπάρχει απαρτία στην Επιτροπή Ρέτζη, οπότε θα ξεκινήσουμε άμεσα τις εργασίες μας. Θέλω να σας προτείνω μια τροποποίηση στην ημίτησια διάταξη. Είχαμε προβλέψει σήμερα το πρωί να συζητήσουμε τον προϋπολογισμό 2020. Μετά τη συνεδρίασή μας συνεδριάζουν συντονιστές, όπου θα πρέπει να παρθούν κάποιες αποφάσεις επί της διαδικασίας. Σας προτείνω λοιπόν το σημείο 4 τη συζήτηση δηλαδή για τον προπολογισμό 2020 να το αφήσουμε για το απόγευμα μετά την ανταλλαγή απόψεων με τη Φιλανδική Προεδρία. Αν δεν έχετε αντίρρηση, δεν βλέπω να υπάρχει αντίρρηση, Υπάρχουν άλλα σχόλια για την ημερήσια διάταξη. Όχι. Παρακαλώ, ο κύριος Ρουζέ. Ναι, συγγνώμη που παρεμβαίνω στο όνομα της ομάδας e ID. Ε, Αξιόριμη Αξιότιμοι είμαι καινούριο εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά δεν είμαι καινούριο στην πολιτική. Εγώ είμαι γκολικός. Και γι' αυτό ακολουθώ τη Μαρίν Λεπέν που είναι η μόνη πολιτικός η οποία ενσαρκώνει ε, το πνεύμα της αντίστασης. Έχω δουλέψει με τον Μισελ Ντεμπρέ, πρωθυπουργό ε, του στρατηγού Ντεγκόλ, έχω εργαστεί ε, με τον Ζακ Σιράκ και κύριε Ρουζέ θέλετε να μας πείτε κάτι για τον κανονισμό Ναι, θέλω να επενθυμίσω τον κανονισμό ε, για τον νόμο Don't. Έμαθα λοιπόν ότι ε, μαθαίνω ότι μεγαλώνουμε όταν σεβόμαστε τη δημοκρατία και όταν σεβόμαστε τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Σας καλώ λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι να σεβαστείτε τον νόμο Don't του Κοινοβουλίου. Έτσι θα σεβαστείτε και τη δημοκρατία, τους κανόνες της, θα σεβαστείτε τους εκατομμύρια ψηφοφόρους μας πως στην Ιταλία και στη Γαλλία έφεραν τη Λέγκα και την ε, ε, εθνική ε, συσπήρωση ε, πρώτους στις χώρες τους και τα εκατομμύρια άλλων ψηφοφόρων και έτσι θα μπορέσετε κι εσείς να δείξετε σεβασμό στους δικούς σας ψηφοφόρους. Μάλιστα, πολύ ωραία σας ακούσαμε να σας πω ότι η Επιτροπή Ρέτζι είναι η οικογένεια των περιφερειών της Ευρώπης αλλά σήμερα είμαστε σε πένθος διότι χάσαμε τον Αντρέ Διόνυσο Μπράτφορντ ο οποίος πέθανε 48 χρονών στις 17 Ιουλίου είχε εκλεγεί σοσιαλιστής ε, ε, ευρωβουλευτής για την περιοχή των Ασόρων ε, και εγώ των Αζόρων και με μεγάλη χαρά τον είχα υποδεχθεί εδώ στην Επιτροπή μας ότι ο Αντρέ ε, ήταν ένας ακούραστος υπερασπιστής των ε, πλέον απομακρυσμένων περιοχών της Ευρώπης δυστυχώς δεν θα είναι πια μαζί μας θέλω να απευθύνω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, στο όνομα όλων σας είμαι βέβαιος προς την οικογένειά του, τους φίλους του στο Σοσιαλιστικό Κόμμα καθώς ε, και τους συνεργάτες του. Υπάρχει ένα βιβλίο, ένα λεύκο με συλληπιτήρια ε, το οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Πορτογάλο συνάδελφο, τον Πέντρο Μάρκες, πριν τηρήσουμε ενό λεπτού γη στη μνήμη του. Ο συνάδελφος έχει το λόγο, παρακαλώ. Thank you so much, Mr. President. Uh, I don't know Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν υπάρχει διερμηνία από τα πορτογαλικά. Θα ήθελα να μιλήσω στα πορτογαλικά, αν γίνεται. Ναι, βεβαίω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για τα λόγια του και όλους τους συναδέλφους για την αλληλεγγύη τους. Ήταν ε, πάρα πολύ μεγάλη απώλεια για μας από την αρχή της θητείας μας. Ε, ο Αντρέ ήταν ε, πράγματι ακούραστος αγωνιστής στις από αποσπασμένες περιοχές. Αγωνίστηκε πάρα πολύ για τις Αζόρες, για την πατρίδα του που την αγαπούσε. Εξαιρετικός άνθρωπος και ουσιαστικά ε, δούλευε στην αντιπροσωπή μας και θα ήταν και ένας μεγάλος ευρωβουλευτής. Είχε μια εξαιρετική οικογένεια. Η γυναίκα του τον αγαπούσε πολύ και αυτός ε, την αγαπούσε. Τέσσερα παιδιά, είχε τη ζωή μπροστά του, αλλά δυστυχώς ε, διακόπη. Με έναν τρόπο πολύ ξαφνικό, φυσικά η πορτογαλική αντιπροσωπεία ε, στεναχωρηθήκε πολύ για αυτή την απώλεια και οι Αζόρες έχασαν ένα μεγάλο πολιτικό αυτής της γενιάς. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και σε διάφορα φόρα αλλά και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης απέτυσε φόρο τιμής σε αυτόν. Ε, εμείς δεσμευόμαστε απέναντι στον Αντρέ και στις Αζόρες ότι θα αγωνιζόμαστε για τις άκροπες απομακρυσμένες περιοχές και για τις αζόρες κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Merci. Je Ευχαριστώ σας προτείνω λοιπόν τον να λεπτού στη μνήμη του. Merci. Comme Όπως γνωρίζετε, θα περάσουμε τώρα ε, στην εκλογή του Προεδρείου, μιας και στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας, είχαμε εκλέξει τον πρώτο αντιπρόεδρο, αλλά σήμερα θα πρέπει να προβούμε στην εκλογή του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου αντιπρόεδρου. Να θυμίσω τα ονόματα των αναπληρωτών που μας νοστοποιήθηκαν στη γραμματεία και ζητώ από... Ναι, παρακαλώ. Θέλετε το λόγο. Η κυρία Κρετού λοιπόν θα αντικατασταθεί από τη Μαρία Γκραπίνη της Σοσιαλιστικής Ομάδας, η κυρία Κρέμ από τον Τόμινο Πεκούλα, η κυρία Σολής Πέρεθ Σουσάνα από τον Μάριος Πέτερς, ο Βίκτορ Ουσπακίτς από την Λογόνς Φαγάντ και για την Γκουε NGL ο Δημήτρης Παπαδημούλης αντικαθιστά τη Μαρτίνα Πίτσελς. Η κυρία Γκεμάν και Αγά στους μη εγγεγραμμένους και ο κύριος Μπόγκοβιτς αντικαθιστέται από τον Σάιλφο Μπούντα δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι αναπληρωτές όχι μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στην ψηφοφορία για τον δεύτερο αντιπρόεδρο. Υπάρχει ε, απαρτία. Θέλω να ζητήσω από τις πολιτικές ομάδες να μας νοστοποιήσουν τους υποψήφιους Παρακαλώ, ναι. Συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. κάτι επί της διαδικασίας. Εμείς ε, θα θέλαμε να αναβληθεί η εκλογή του τετάρτου αντιπροέδρου για το απόγευμα ή ακόμα καλύτερα για τον Σεπτέμβριο. Θα ήθελα λοιπόν να αποφασίσουν οι συνάδελφοι. Πολύ ωραία. Ανακοινώνω την ψηφοφορία για το δεύτερο αντιπρόεδρο. Υπάρχει μία υποψηφιότητα και θα δώσω το λόγο στην ομάδα Renew. Σας ευχαριστώ για το λόγο. Κυρίες και κύριοι, είναι τιμή μου να σας παρουσιάσω τον κύριο Κριστιαν Γκίνεα που κάθεται δεξιά μου και να σας τον παρουσιάσω ως τον υποψηφιό μας για την δεύτερη αντιπροεδρία της Επιτροπής Ρέτζη. Ο κύριος Γκίνεα έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρο τη διαδρομία του. Εργαζόμενος για τις ευρωπαϊκές ιδέε ως δημοσιογράφος, ε, έχει ιδρύσει και ένα επιτυχές think tank στη χώρα του. Επίσης, εργάστηκε ως υπουργού ε, για τις ευρωπαϊκές ε, υποθέσεις στη Ρουμανία. Πιστεύουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να υποστηρίξει την Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Ωραία. Θα πρέπει να συγκατατεθεί και ο κύριος Γκίνα, συμφωνείτε. Πολύ ωραία. Διαπιστώνω ότι έχετε συμπληρώσει και τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων καθώς και την δήλωση σε σχέση με τον κώδικα δεντολογίας και θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματος ε, της ομάδας CCR θα ήθελα να καταλάβω αν η πρόταση έγινε πριν ε, από το να μας ε, πείτε για τις εκλογές του Δευτερού του Προέδρου, δηλαδή το θέμα της αναβολής του Τέταρτου του Προέδρου. Πριν να ψηφίσουμε για δεύτερο και τρίτο αντιπρόεδρο, να ξέρουμε αν είμαστε ε, ενώπιον μιας ε, ήδη προδιαγεγραμμένης ε, πλειοψηφίας. Εγώ θεωρώ ότι είναι περίγραπτο να αποκλείονται κάποιες ομάδες. Έτσι λοιπόν αν έχει διποφασιστεί ότι όλοι οι κανόνες και η δυνατότητα να συμπεριφερθούμε κατάλληλα σε αυτή την επιτροπή απέναντι στις διάφορες ομάδες καταπατούνται, αν είναι έτσι να το σημειώσουμε, αλλά πρέπει να το ξέρουμε πριν από την ψηφοφορία για δεύτερο και τρίτο αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ. Très bien. Je Πολύ ωραία. Το ανακοίνωσα όταν ξεκίνησε τις εργασίες της Επιτροπής μας. Σήμερα το πρωί θα προχωρήσουμε στην εκλογή του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου Αντιπροέδρου. Έχουμε καταγράψει μία υποψηφιότητα, μία και μόνη υποψηφιότητα για τον δεύτερο Αντιπρόεδρο από την ομάδα Ρινιού, τον συνάδελφο Γκίνεα. Δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες, έτσι λοιπόν ε, σας ζητώ διαβοής να ψηφίσετε αν ε, θέλετε να εκλεγεί ο κύριος Γκίνεα. Και θα τον καλέσω εδώ στο βήμα να καθίσει δίπλα από τον συνάδελφο Έτμαν. Selon la même procédure, nous allons... Με την ίδια διαδικασία θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία για τον τρίτο αντιπρόεδρο. Il n'y a pas d'autres suppléants. Δεν υπάρχουν άλλοι αναπληρωτές. Έτσι λοιπόν, ζητώ από τους υποψηφίους να αυτοπερισιαστούν για τους σοσιαλιστές, κύριο Κοτσελίνο. Προτείνουμε τον συνάδελφο Αντριάν Τράγκο ω τρίτο αντιπρόεδρο. Προέρχεται από την Ρουμανική Αντιπροσωπεία. Notre collègue Dragos donne-t-il son... Συμφωνεί ο κύριο Δράγκος. Ναι, συμφωνώ. έχετε δεόντως συμπληρώσει και την δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα, επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκλογή διαβοής. Πρόεδρε, εγώ ήθελα να ψηφίσουμε και όχι να εκλεγεί διαβοή αν είναι δυνατόν. Καθώς υπάρχει μία και μόνη υποψηφιότητα, η εκλογή διαβοής επιβάλλεται. Σας ευχαριστώ. Μπορείτε να έρθετε στο βήμα. un rappel au règlement. Sì, solo per... Πρόεδρε, θα ήθελα να καταλάβω την ε, αρχή που διέπει την ψηφοφορία. Γιατί στην Επιτροπή Επασχόληση, ε, παραδείγματο χάρη, ψηφίσαμε για ένα και μόνο υποψήφιο που ήταν ε, και για τον πρόεδρο και κάθε φορά απορρίφθηκε αυτός ο υποψήφιος. Ενώ τώρα μαθαίνω ότι αν υπάρχει ένας και μόνο υποψήφιος, εκλέγεται διαβοής. Δεν χρειάζεται η Επιτροπή ε, Ρέτζι να ακολουθήσει το τι κάνει η Ταδίδιν Επιτροπή. Εμείς ακολουθούμε τους δικού μα κανόνες. Είναι στην αρμοδιότητα του Πρόεδρου να αποφασίσει. Και πιστεύω ότι όταν δεν υπάρχει παρά μόνο μία υποψηφιότητα, δεν χρειάζεται να περιπλέκουμε τα πράγματα. Και η εκλογή διαβοή είναι δυνατή. Να περάσουμε λοιπόν στην εκλογή του τέταρτου αντιπροέδρου. Υπάρχουν υποψηφιότητες. Ένα διαδικαστικό σημείο. Νοβάκοφ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα για πρώτη φορά να παρουσιάσω μια κυρία για να έχουμε και μια ισορροπία σε ό,τι αφορά το φύλλο. Θα ήθελα λοιπόν να παρουσιάσω την Ιζαμπέλ Μπέχουμερ που πιστεύω ότι πληρεί όλες τις απαραίτητες ε, προϋποθέσεις ε, για να γίνει αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, Ρέτζη. Ήδη έχει αποδείξει τις ικανότητες της για να εργάζεται στην περιφερειακή ανάπτυξη. Προέρχεται από την Ισπανία. Έτσι λοιπόν ταπεινά ζητώ από όλους τους συναδέλφους να την υπερψηφίσουν. Très bien. Madame Isabelle η κυρία Ιζαμπέλ ε, Μπεν συμφωνείτε. Ναι, ναι, τα έχουμε. Ευχαριστώ. Έχετε κι εσείς πληρώσει ιδεόδος τη δήλωση συμφερόντων καθώς ε, και τη δήλωση για την κωδίκα δεντολογίας. Υπάρχουν ε, άλλες υποψηφιότητες. Παρακαλώ. καθώς ε, πρόκειται για κάποια κριτήρια που πρέπει να πληρούνται, καθώς ε, έλειπε και η ποσόστοση του γυναικείου φύλου, όπως ε, ήδη εκφράστηκε την περσμένη φορά, η ομάδα ID προτείνει εκ νέου πάλι μια κυρία ως υποψήφια, την κυρία Φρασένσκα Ντονάτο, η οποία είναι σε θέση οπωσδήποτε να πληρεί τη θέση της Αντιπρόεδρου προέρχεται από τη Σικελία. Είναι μια περιοχή συνοχής, μακρινή και συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά και πολιτικά και υλικά για να ε, μπορέσει να λάβει το ρόλο της τέταρτης αντιπροέδρου. Κυρία Φραντσέσκα Ντονάτο, συμφωνείτε? Τέλεια. Έχετε κι εσείς συμπληρώσει δόντω την δήλωση συμφερόντων και έχουμε δύο υποψήφιους, δύο υποψήφιες. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Όχι. Σας προτείνω λοιπόν να προχωρήσουμε σε μια ψηφοφορία ηλεκτρονική. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων ε, να ελέγξετε αν έχετε τις κάρτες σας και θα είναι μυστική η ψηφοφορία. Λοιπόν.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 Ιζαμπέλ Μπεχομέα, πατούν το πράσινο κουμπί. Όσοι θέλουν να ψηφίσουν την υποψήφια της ομάδας ID, την κυρία Ντονάτο, πατούν το κόκκινο κουμπί. Κανονικά αποχές δεν υπάρχουν. Βεβαίως, εάν κάποιος θέλει να απόσχει, μπορεί να πατήσει το άσπρο κουμπί. Είναι σαφή τα πράγματα για όλους. Είναι μυστική η ψηφοφορία αυτή, επαναλαμβάνω. Άρχεται η ψηφοφορία. Il y a PPE de trop. Περισσεύουν δύο βουλευτές του ΕΛΚ. Οπότε θα ήθελα να σας ζητήσω, να ζητήσω από δύο αναπληρωματικά μέλη να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Ωραία. πέρα της ψηφοφορίας και εδώ βλέπετε το αποτέλεσμα 26 ψήφοι υπέρ της Ιζαμπέλ Μπεχουμέα 8 ψήφοι για τη συνάδελφο την κυρία Ντονάτο. Η Ισαμπέλ Μπεχουμέα λοιπόν εκλέγεται ως τέταρτη αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας. Και θα ήθελα να τη ζητήσω να έρθει και αυτή εδώ στο Προεδρείο. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τις πολιτικές ομάδες που έκαναν ε, αυτή την προσπάθεια ε, να σεβαστούν ε, την ισορροπία στο Προεδρείο και σε γεωγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο εκπροσώπησης των δύο φύλων. Ε, είναι πλήρες πλέον το Προεδρείο και μπορούμε πλέον να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Σήμερα το απόγευμα θα έχουμε μια σημαντική συνάντηση με την Φιλανδική Προεδρία και στη συνέχεια θα έχουμε τη συζήτηση για τον προπολογισμό του 2020. Σε λίγο θα συναντήσουμε τους συντονιστές, ε, θα έχουμε συνάντηση συντονιστών, εν πάση ε, όταν θα διακόψουμε για το καλοκαίρι, πρέπει να σας πω ότι μετά θα έχουμε εξαιρετικά εντατικούς ρυθμούς, μιας και θα χρειαστεί δίχως άλλο να ξεκινήσουμε τον τρίλογο, τον τριμερή διάλογο για τα ταμεία που αφορούν ε, τα, γενικό κανονισμό αλλά και το Ταμείο Συνοχής. Ε, πολύ σημαντικό το διακύβευμα για την Επιτροπή Ρέτζη και επιστολή την προσοχή σας στη μάχη που θα πρέπει να δοθεί με το Συμβούλιο για τον προπολογισμό. Είναι κεφαλαιόντως σημασία σε αυτή η μάχη και με ελάχιστε εξαιρέσει φαντάζομαι ότι όλοι σας εδώ ε, θέλετε να υποστηριχθεί η περιφερειακή πολιτική. Και στη δική σας χώρα πρέπει να δώσετε τη μάχη. Πρέπει να φτάσει το μήνυμα και στις κυβερνήσεις σας ότι η συνοχή πρέπει να έχει επαρκή κονδύλια, επαρκή προπολογισμό για να μπορεί να υπάρξει ένας δυναμικός προγραμματισμός και να μην οπισθοδρομήσουμε. Είναι λοιπόν κρίσιμη αυτή η μάχη. Η Επιτροπή Ρέτζη θα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης και θα ήθελα σήμερα το απόγευμα ε, στην συνάντηση με την Φιλανδική Προεδρία να φανούμε στο ύψος των περιστάσεων, διότι αυτή η Προεδρία θα είναι κρίσιμη ε, για την προπαρασκευή των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πολιτισμό οικονομικό πλαίσιο, ενδεχομένως να ολοκληρωθούν και επί Φιλανδικής Προεδρίας, ε, αν και αυτό θα είναι κάπως δύσκολο. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν το απόγευμα. Ζητώ από τους συντονιστές να μείνουν στην αίθουσα και δίνω ραντεβού στα μέλη για να ξεκινήσουμε εκ νέου τις εργασίες μας το απόγευμα με την Φιλανδική Προεδρία στις 3. Ευχαριστή γενικά και τις δερμηνείς ο Πρόεδρος.